θα προσαρτηθεί ο κατάλογος στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις που θα γερθούν, θεωρούνται αυτοί οι διορισμοί ότι έχουν εγκριθεί από την Ολομέλεια. Ερχόμαστε τώρα στις δήλωσεις αντιπροέδρου της Κομισιόν και υπά του εκπροσώπου για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σε σχέση με την κατάσταση στην Αίγυπτο. Δίνω το λόγο στον εκπροσωπούντα την κυρία Άστον, τον κύριο Μαυρογιάννη. Κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι Αιγύπτιοι μπόρεσαν να εκφράσουν ελεύθερα την γνώμη τους, τη θέση τους για να επιλέξουν το άτομο το οποίο είναι ο φορέας των ελπίδων τους και των προσδοκιών τους. Το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της 25ης Ιουνίου έχει επενέσει την ειρηνική διανέργεια των εκλογών που είναι ένα σημαντικό βήμα μέσα στην δημοκρατική μετάβαση της Αιγύπτου. Ο πρόεδρος Φαν Ρομπόι, ο πρόεδρος Μπαρόσο, η Καθρίν Άστον και πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συγχαρεί τους Αιγυπτίους και τον νέο πρόεδρο της Αιγύπτου για αυτή τη σημαντική ιστορική αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή <clears throat> ε, Ένωση μέσω της ε, εκλογικής αποστολής παρακολούθησής της και οι διάφορες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν αναφέρει κάποια συστηματική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μπορούσε να έχει αλλάξει το αποτέλεσμα των εκλογών. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την ε, παρακολούθηση των εκλογών και συντονισμό αυτής της διεθνούς παρουσίας στο Κάιρο. Είναι υψής της σημασίας ότι με την ηγεσία του Πρόεδρου Μόρση όλοι οι Αιγύπτιοι θα μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως των δημοκρατικών ελευθεριών τους και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και αυτό να, ότι θα μπορέσει να εξασφαλίσει την ανάτηση μιας ανεξάρτητης και ενεργού ε, κοινωνίας των πολιτών. Έχουμε τονίσει λοιπόν <clears throat> ότι χαιρόμαστε για τη θέληση του κυρίου Μόρση να τηρήσει όλες τις διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Αίγυπτος. και η σταθερότητα όλης της περιοχής αυτής που είναι η δική μας γειτονιά είναι ένας κοινό στόχος και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Αίγυπτο. Η συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ της Αιγύπτου διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο. Το ανώτατο δικαστήριο των ε, ενόπλων δυνάμεων έχει εξασφαλίσει ότι θα παραμείνει ενισχύ αυτή η συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ και θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική της Αιγύπτου. Οι αρχές της Αιγύπτου επίσης θέλουμε να διαδραματίσουν ένα επικοδομητικό ρόλο για να αντιμετωπιστούν όλες οι προκλήσεις της περιοχής και αυτό έχει να κάνει επίσης και με τη συμφιλίωση των φατριών στην Παλαιστίνη. Η διαδικασία μετάβαση πρέπει να συνεχίσει και ο δρόμο για μια εδρεωμένη και βιώσιμη δημοκρατία η οποία θα ανταποκριθεί στις προσδοκίε και τι επιθυμίε των Αιγυπτίων. Αυτό είναι ένα μακρό δρόμο που θα πρέπει να διατρέξουμε, αλλά δεν υπάρχει επιστροφή για την Αίγυπτο, έχει ήδη δεσμευτεί προ αυτήν την κατεύθυνση. Στι 27 Ιουνίου η απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου των Ενόπλων Δυνάμεων, η απόφαση αυτή να διαλυθεί η κάτω βουλή στην Αίγυπτο είναι κάτι το ανησυχητικό, διότι με αυτό το διάταγμα το Ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων έχει αναλάβει νομοθετικές εξουσίες και έχει σε σημαντικό βαθμό περιορίσει τις εξουσίες του δημοκρατικά εκλεγμένου Πρόεδρου. Το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της 25ης Ιουνίου εξέφρασε τις σοβαρές ανησυχίες του σε σχέση με αυτές τις εξελίξεις. Η, και αντιπρόεδρος κάθε άστον παραμένει σε στενή επαφή με τι αρχέ τη Αιγύπτου. Όλε οι εμπλεκόμενε πλευρέ θα πρέπει να βρουν μια λύση η οποία επιτρέπει την πλήρη μεταφορά τη εξουσία σε δημοκρατικά εκλεγμένου πολιτικού φορεί, μη στρατιωτικού φορείς, το ταχύτερο δυνατόν. <clears throat> Μέσα στα πλαίσια αυτά, η δεδηλωμένη πρόθεση του κυρίου Μόρση να έχει ένα κυβερνητικό σχηματισμό που εκπροσωπεί όλες τις δυνάμεις της Αιγύπτου, αυτό είναι κάτι το πολυθετικό. Μπορεί με τον τρόπο αυτό να συμβάλλει σημαντικά στο να προκύψει μια εθνική συνένεση η οποία είναι απαραίτητη για την διάρκεια της λεπτής αυτής φάσης μετάβασης. Στους επόμενους μήνες θα υπάρξει σημαντικός αντίκτυπος για το μέλλον της Αιγύπτου, πρέπει να υπάρξει το νέο σύνταγμα και θα πρέπει να υπάρξει κατά πάσα πιθανότητα και μια νέα εκλογική διαδικασία. Ένα βασικό στοιχείο αυτής της, μεταβατικής, της δημοκρατικής μετάβασης είναι το να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει δυνατότητα όλων να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή χωρίς να υπάρχει το φάσμα του φόβου, ανεξάρτητα από την πολιτική του τοποθέτηση, το φύλλο, τη θρησκεία ή τις πεπιθήσεις. Από την ίδια τη φύση του, το Σύνταγμα είναι ένα θεμελιακό σύμφωνο, το οποίο πρέπει να είναι συνενετικό και περιεκτικό για να μπορεί να είναι ένα ανθεκτικό σημείο αναφοράς για όλους τους πολίτες. Αναμένουμε λοιπόν ότι οι διατάξεις, οι πρόνοιες του νέου αυτού συντάγματος θα προστατεύσουν καταρχήν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ε, ελευθερίες όλων των πολιτών. Δεύτερον, ότι θα θέσουν τον στρατό και την αστυνομία κάτω από τον έλεγχο δημοκρατικά εκλεγμένων πολιτικών αρχών <clears throat> και τρέτον θα εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Η Αίγυπτος μπορεί να βασιστεί στην στεναρή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσει τα πολύπλοκα αυτά προβλήματα και τις κοινωνικονομικές προκλήσεις ενώπιών της. Προσβλέπουμε λοιπόν σε μια στενή και καρποφόρα συνεργασία με τον νέο πρόεδρο Μόση και με τη μελλοντική κυβέρνηση της Αιγύπτου, στοχεύοντας να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις διμερείς μας σχέσεις Δία να επιτύχουμε κάτι τέτοιο, ο διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αιγύπτου θα πρέπει να επαναληφθεί το ταχύτερο δυνατό. Μία από τις προτεραιότητές μας είναι ότι στο νέο σχέδιο δράσης που θα πρέπει να συντάξουμε να αντικατοπτρίζονται οι στόχοι της πολιτικής γειτονίας όπως καθοριστήκαν τον Μάρτιο και τον Μάιο του 2011 σε αντίστοιχες ανακοινώσεις. Η ειδική μονάδα λοιπόν για την Αίγυπτο που θα συγκροτηθεί αυτό το φθινόπωρο θα είναι μια ευκαιρία να καταδείξουμε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συνέχιση της ε, δημοκρατικής μετάβασης στην Αίγυπτο. Η πάτη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Κομισιόν θα θέλει να ε, χαιρετήσει την συνεισφορά όλων σε αυτή την ειδική μονάδα για την Αίγυπτο. Αλλά σε τελική ανάλυση η ευθύνη για το μέλλον της Αιγύπτου, για τη δημοκρατική αυτή μετάβαση βρίσκεται στα χέρια των Αιγυπτίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θα συνεχίζει να πράττει ό,τι είναι δυνατόν για να τους ενισχύσει και να τους βοηθήσει να επιτύχουν στο σημαντικό αυτό εγχείρημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μαυρογιάννη. Ακολουθούν οι ομιλητέ εξ των ομάδων. Ο κύριο Πέτριν για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Αίγυπτο εξέλεγε ένα πρόεδρο σε εκλογέ χωρίς βία και αυτό είναι θετικό και αξιοσημείωτο για την Αίγυπτο. Η ομάδα του ΕΛΚ εύχεται στον νέο πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Μοχάμετ Μούση, καλή επιτυχία και ευχόμαστε να έχουμε καλή συνεργασία. Οι πρώτες δηλώσεις του νέου Προέδρου είναι ενθαρρυντικές. Αυτά τα οποία είπε σε σχέση με τη δουλειά του όσον αφορά τις μειονότητες, χριστιανούς, κόπτες είναι υπόδειγμα για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο. Ο πρόεδρος Μουσή είπε πως θα μπορούσε αντιπρόεδρος να είναι ένας κόπτης και θα έκανε άρα κάτι το οποίο θα έρχονταν σε με άλλες δηλώσεις από τον αραβικό κόσμο, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο είπε ο μεγάλος μουφτής της Σαουδικής Αραβίας, που απορώ ε, για το ότι δεν βρήκε μεγαλύτερη δημοσιότητα γιατί είπε πως στην Αραβική Χερσόνησο πρέπει να καταστραφούν όλες οι εκκλησίες και να μην χτιστούν άλλες. Και αν ακολουθήσει άλλο δρόμο η Αίγυπτος και πει πως μπορούν να συνεπάρξουν θρησκεία και πολιτική θα έχουμε ένα νέο παράδειγμα για το ότι η Ισλαμική πίστη και η πολιτική μπορούν να συνεπάρξουν. Και το λέω ξεκάθαρα ως χριστιανός. Δεν υπάρχει χριστιανική πολιτική, αλλά υπάρχει πολιτική χριστιανικής ευθύνης. Και αντιστοίχως δεν μπορεί να υπάρξει μουσουλμανική πολιτική, αλλά μπορεί να υπάρξει μια πολιτική με αφετηρία την μουσουλμανική πίστη. Δηλαδή με τον άνθρωπο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στο κέντρο της, κάτι με το οποίο νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Ένα θετικό μήνυμα είναι επίσης πως ο πρόεδρος Μούση είπε πως θα τηρήσει τις διεθνείς συμφωνίες και άρα τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ ε, των πρόεδρων Σαντάτ και Μπεγκίν και κύριε Υπουργέ, κύριε Μαυρογιάννη θα σας ήμουν ε, ευγνώμων ε, εάν ε, θα μπορούσατε να ζητήσετε να μην προσμετρηθεί αυτό στον χρόνο μου. Τέλος για το Ισραήλ βεβαίως ζήτησε να σταματήσει η πολιτική των ε, επικισμών. Επίσης, κάτι τελευταίο. Δεν είναι δυνατόν μη κυβερνητικέ οργανώσεις και διεθνείς, ε, διεθνή ιδρύματα όπως το Ίδρυμα Κόναντ Αντενάουρ να σέρνονται στα δικαστήρια για υποτιθέμενη παράνομη δραστηριότητα. Πρέπει να αντιληφθούν πως θα πρέπει να σταματήσει αυτή η δίκη. Οι Αιγυπτιακές αρχές θα πρέπει να μπορούν να δουν ελεύθερα άνθρωποι από την Ευρώπη, από ολόκληρο τον κόσμο, από την κοινωνία των πολιτών για να μπορέσει να συνεισφέρει και η κοινωνία των πολιτών στην δημοκρατία και την ελληνική εξέλιξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μπορούμε να πούμε ότι επιτέλους η επίσημη ανακοίνωση της ε, ανάγκης των καθηκόντων του ε, κ. Μόρση ε, δείχνει μια πρώτη φάση των πολιτικών εξελίξεων στην Αίγυπτο και αυτό δεν ήταν δεδομένο πριν από αυτή τη διακήρυξη και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι μέρες αυτές είχαν συγκλονιστεί από δύο αποφάσεις του Δημοτικού Δικαστηρίου ε, στην πρώτη αποφάση θεώρησε μη συνταγματικό την Ένωση της Πολιτικής Απομόνωσης που θεωρούσε ότι δεν είναι νόμιμη ε, η υποψηφιότητα του σαφή στι προεδρικέ εκλογέ και δεύτερο θεώρησε μη συνταγματική τον εκλογικό νόμο για τι κοινοβουλευτικέ εκλογέ και βάσει αυτού διέλυσε το Κοινοβούλιο. Και αυτό θα μπορούσε να έχει συνέπειε και όσον αφορά και την συνταγματική συνέλευση. Περιέβρισκαν τα πράγματα και οι τροπολογίες όσον αφορά τη συνταγματική δήλωση που ακυρώθηκε από το Νότιο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδυναμώνουν αυτά τα μέτρα της εξουσίας του Προέδρου και καταργούν την νομοθετική εξουσία και αυτόνομη ε, μέχρι την έγκριση νέου συντάγματος. Στην πρώτη ομιλία σαν Πρόεδρος, ο Μόρση ε, έστειλε ένα μήνυμα ενότητας και συμφιλίωσης προσπαθώντας να καθησυχάσει τις διάφορες συνιστώσεις της, Ευρωπαϊ... της Αιγυπτιακής κοινωνίας. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική θεωρήσε ότι θα είναι πιστός στις διεθνές υποχρεώσεις που έχουν αναλυφθεί. Θα δούμε κατά πόσο θα ακολουθήσουν οι πράξεις τα λόγια. Εν πάση περιπτώσει, μετά από μια περίοδο άκρα αβεβαιότητα και ασταθία, η, η εκλογή του νέου Προέδρου θα μπορούσε επιτέλου να ανοίξει μια νέα φάση που μπορεί από τη μια πλευρά να οδηγήσει την Αίγυπτο γρήγορα προς εφαρμογή της, της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων και μετά θα μπορούσε να οδηγήσει τις προσπάθειες για ανάκαμψη της οικονομίας και να διορθωθεί και να αποκατασταθεί η χρηματοσυντική κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει σαφής ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και μέσω της Task Force της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Αιγύπτου. Θα πρέπει η Ευρώπη να είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον νέο Πρόεδρο για να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις, για να υποστηρίξει και να δείξει σε καλό τέρμα τη διαδικασία της δημοκρατικής μετάβασης και για να ξεπεραστεί η οικονομική και χρηματοστηρική κρίση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο η σταθερότητα της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παντσέρη. Η κυρία Σάκη για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο λαός της Αιγύπτου μαζί με πολλούς άλλους λαούς έχουν γιορτάσει την ιστορική εκλογή του πρώτου ελεύθερα εκλεγμένου Προέδρου που δεν είναι και στρατιωτικό ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Το ανώτατο Συμβούλιο όμως των Ενόπλων Δυνάμεων έχει διαλύσει το Κοινοβούλιο και έχει αυξήσει τις εξουσίες του παρεμβαίνοντας και στην νομοθετική και εκτελεστική εξουσία. Εμείς θα πρέπει μαζί με του Αιγυπτίου να κατανοήσουμε ότι υπάρχει πολλή δρόμο για να διατρέξουμε μέχρι ότου η Αίγυπτο είναι πλήρω δημοκρατική. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να αλλάξει ο πρόεδρο Μόρση τη στιγμή που τα βασικά στοιχεία μια δημοκρατία, όπω είναι η διαίρεση των εξουσιών, ο διαχωρισμό των εξουσιών και το κράτο δικαίου, δεν ισχύουν. Συνεχίζεται ακόμα να υπάρχει στρατιωτική εξουσία στην Αίγυπτο. Ζητήσαμε να καταργηθεί άμεσα ο στρατιωτικό νόμο και τα στρατοδικεία. Είναι απαράδεκτα το να είναι τόσα πολλά άτομα στι φυλακέ για πολιτικά αδικήμενα και ακόμα είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο να καταδικάζονται από στρατοδικεία χωρί δίκαια δίκη. Μόνο αν σταματήσουν αυτέ οι δίκε σε στρατοδικεία, σταματήσουν, μπορεί να θεωρεί η Αίγυπτο ότι είναι κράτο δικαίου και αν γίνουν σεβαστά τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη κάθε άστον θα πρέπει να πιέσει την Αίγυπτο να σεβαστεί τα δικαιώματα όλων των Αιγύπτιων. Οι εκλογέ θα πρέπει να οδηγήσουν σε ένα κοινοβούλιο το οποίο είναι πραγματικά αντιπροσωπευτικό και το οποίο θα έχει πραγματικέ νομοθετικέ εξουσίε. Εμεί θα δώσουμε το ωφέλιμα τη αμφιβολία στον πρόεδρο Μόρση. Αλλά θέλουμε να τονίσουμε ότι οι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά έναντι μεγαλύτερου σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και τη δημοκρατική διαδικασία και επίση δικαιωμάτων των γυναικών, εξακολουθεί να ισχύει αυτή η αρχή. Όλε οι νέε εξουσίε στην Αίγυπτο θα κρυθούν από τι πράξει του. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε για αυτή τη δύσκολη αλλά σημαντική διαδικασία μετάβαση όταν υπάρχουν πραγματικά βελτιώσει που μπορούν να θεωρηθούν μια πραγματική καμπή, μια επανάσταση, μια μετάβαση από την ε, καταπίεση στην ελευθερία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σάκε η κυρία Μπεναράπ Ατού για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά την πτώση του Μουμπάρακ το Φεβρουάριο του 2011 η Αίγυπτος διοικείται από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων που πήρε την εξουσία να νομοθετεί και να συντάσει το Σύνταγμα. Και γι' αυτό ανησύχησε το, η χώρα. Και αυτό 24 Ιουνίου που πέρασε ο Μοχάμετ Μόρσε, του, των αδελφών μουσουλμάνων, εξελέγει για πολλούς ε, Αιγυπτίους αυτή η εκλογή ε, ίσως ε, να, να υποβαθμίζει κάπως την, την ομοθεσία. Λοιπόν, θα μπορούσαν οι γυναίκες ναι, κανονικά να δια... χωρίς συμφωνία των συζύγων θα μπορούσαν να παίρνουν διαζύγιο και θα μπορούσαν οι γυναίκε λοιπόν θα πρέπει να ακουστούν Και τώρα στι διεκδικήσει που έχουν, χωρί αυτέ η δημοκρατία στην Αίγυπτο δεν θα είναι δυνατή. Λοιπόν, αυτό λοιπόν απαιτούν να υπάρξει η χάρτα των ε, δικαιωμάτων των γυναικών στην Αίγυπτο που κατατίστηκε υπογράφει πάνω από χίλιε γυναίκε και νεκρήθη από 1,5 εκατομμύριο Αιγύπτιου πολίτε, άνδρε και γυναίκε. Λοιπόν, αυτό το έγγραφο καθεγιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα όπω το δικαίωμα τη συμμετοχή στην πολιτική ζωή, στην οικονομική ζωή, την εκπροσώπηση εντό τη κυβέρνηση και την ισότητα αντι του νόμου. Η Αιγυπτιακή δικαιοσύνη θα πρέπει να προστατεύει τι γυναίκε κατά κάθε παραβίαση, κάθε μορφή βία. Ε, θα πρέπει απολύτω να υποστηρίξουμε αυτέ τι διεκδικήσει, οι οποίε είναι θεμητέ και νόμιμε. Η κυρία Άστον θα το κάνει. Ε, ποια μέτρα ε, έχει υπόψη τη να ε, θέση για να συνοδεύσει στη δημοκρατικό δρόμο την Αιγύπτιο. Πώ πάντα αποκριθούμε στο φόβο των γυναικών εμεί οι Ευρωπαίοι που φοβούνται ότι οι Ισλαμιστέ θα καταβατήσουν τα δικαιώματά του και την διακόπτη την ομιλήτρια, Πρόεδρο. Πατού. Συγχωρείτε, κύριε συνάδελφε. Ε, Ούτω ή άλλω είχε τελειώσει ο χρόνος σας αλλά προσπάθησα να σας κάνω και ένα νόημα να μιλάτε λίγο πιο σιγά για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και οι ε, έπρεπε είτε να σα κάνω νόημα είτε να σας αφαιρέσω το λόγο αλλά ούτω ή άλλω είχε τελειώσει ο χρόνο. σας ο κύριο Τάνοκ για ένα λεπτό Έχουμε λοιπόν τον πρώτο δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο μετά την εποχή Μπάρακ και βεβαίως θα πρέπει ο Μούση να τηρήσει δύο βασικές υποσχέσεις. Πρώτα απ' όλα την ε, ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ και βεβαίως να δεσμευτεί για να βρεθεί μία λύση για το άραβο-ισραηλινό ζήτημα με μία λύση δύο κρατών. Επίσης βεβαίως πρέπει να σε δει τι θα κάνει με την κοπτική μειονότητα και να την προστατεύσει από τις διώξεις που υφίσταται από σαλαφιστές ακραίους. Οπότε καλωσορίζω την δεσμευσή του να συμπεριλάβει γυναίκες και χριστιανούς στην κυβέρνησή του και πρέπει αυτή τη στιγμή να αποστασιοποιηθούν η οι αδελφοί μουσουλμάνοι από τα ακραία στοιχεία που θέλουν να επιβάλλουν σε ουδικού τύπου κυβέρνηση που θα οδηγήσει σε απομόνωση την Αίγυπτο και πιθανώς σε μαζική έξοδο χριστιανών και κατάρρευση της Αιγυπτιακής οικονομίας. Σας ευχαριστούμε. κυρία Ματίας, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι η εκλογή του Πρόεδρου Μωάμεντ Μόρση μετά από την εποχή του Μουμπάρακ είναι μια μεγάλη επιτυχία. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε ψευδεστήσεις γιατί αυτές οι προεδρικές εκλογές δεν επηρεάζουν με κανένα τρόπο τη διαδικασία μετάβασης στην Αίγυπτο. Όπως αναφέρθηκε υπήρξε η διάλυση του Κοινοβουλίου 10 μέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές και τονίζει την ύπαρξη κινδύνων. Η εξουσία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι Υπερβολικοί Έχουν εκτελεστική εξουσία, έχουν νομοθετική εξουσία, περιορίζουν την λειτουργία του Πρόεδρου και φυσικά αυτοί θα αποφασίσουν ποιε αλλαγέ θα υπάρξουν στο Σύνταγμα. Όλα αυτά μα ανησυχούν και θα πρέπει να θέσουμε ερωτήματα στου εαυτού μα. Η Αίγυπτος κινδυνεύει να παραμείνει στα χέρια της στρατιωτικής εξουσίας. Όταν διαλύεται ένα κοινοβούλιο ή όταν δεν είναι πραγματικά εκλεγμένο, τότε αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πλήγμα στη δημοκρατία. Πρέπει εμείς λοιπόν ως Ευρωπαίοι να υποστηρίξουμε όλες τις προτάσεις για την δημοκρατική αλλαγή που προτείνει η αντιπολίτευση και να υποστηρίξουμε την ανάγκη να υπάρξει ένα δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κύριος Μπέλντερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είχα επαφές ε, χθε το βράδυ με χριστιανούς στην Αίγυπτο και μάθα πως ανησυχούν πάρα πολύ για την κατάσταση στην πατρίδα του. Τα ε, ενισχυτικέ ε, δηλώσει και χειρονομίε του νέου πρόεδρου, ο οποίος είναι αδελφός μουσουλμάνος του κ. Μουχάμεντ Μόρση, δεν τους καθησυχάζουν. Μην ξεχνάμε πως από την πτώση του Μουμπάρακ ήδη οι αδελφοί μουσουλμάνοι σε κρίσιμες στιγμές έχουν παραβιάσει τρεις φορές παραβεί υποσχέσεις τους. Οπότε θα πρέπει η ύπατη εκπρόσωπος να τονίσει το θέμα της χριστιανικής μειονότητας στις επαφές της με τις Αιγυπτιακές αρχές. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να τεθεί ενώπιον του Καΐρου είναι οι παγωμένες σχέσεις με τη γειτονική χώρα, το Ισραήλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τονίσει την ηγεσία του Αιγυπτιακού στρατού πως πρέπει να αποκατασταθεί ο έλεγχος των συνόρων τους με το Ισραήλ στη χερσόνησο του Σινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπέλτερ. Για ένα λεπτό ο κύριος Όμπερμαϊρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι χριστιανοί στην Αίγυπτο φοβούνται ότι με την εκλογή του νέου Προέδρου, ο οποίος εκπροσωπεί τους αδερφούς μουσουλμάνους, ανοίγει ο δρόμος για ένα Ισλαμικό κράτος που θα είναι κόλαση για τους κόπτες. Οι κόπτες φτάνουν περίπου το 20% του πληθυσμού στην Αίγυπτο, μιλάμε δηλαδή για 10 εκατομμύρια περίπου άτομα, που δεν είναι πάντα όλοι ανοιχτά έτοιμοι να αναγνωρίσουν αυτό το, το του. Υπάρχει ο κίνδυνος σε ένα Ισλαμικό καθεστώς να είναι άτομα χωρίς κανένα δικαίωμα. Η Ισλαμική παρουσία δεν είναι καινούρια στην περιοχή αυτή. Ήτανε κάτι το οποίο είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν ως παράταξη, αλλά τώρα κινδυνεύει να γίνει μια κυβέρνηση. Δεν υπάρχει πια κανένα ίχνος από την Αραβική Άνοιξη. Η κυρία Άστον θα πρέπει να αξιολογήσει αμέσως την κατάσταση των χριστιανών στην Αίγυπτο και να τονίσει την ανάγκη να τηρηθούν και να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Όμπερ Ακολουθεί η σειρά των άλλων ομιλητών από τι πολιτικέ ομάδε. Δύο λεπτά, κύριο Μίλαν μόνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ χαίρο, χαιρετίζω το γεγονό ότι οι εκλογέ προεδρικέ στην Αίγυπτο έγιναν χωρί μείζωνα προβλήματα και, είχαν, και έγιναν δεκτά τα αποτελέσματά του. Αλλά είναι σαφέ ότι οι εκλογέ αυτέ και οι ε, απρόπτε αποφάσει που λήφθησαν από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων στην Αίγυπτο καταδεικνύουν ότι στην πραγματικότητα υπάρχει διτή εξουσία στην Αίγυπτο. Είναι δύσκολε στιγμές είναι απαραίτητο οι δύο αυτοί πόλοι, τα δύο αυτά κέντρα εξουσίας να βρεθούν σε διάλογο και συνεργασία στο τωρινό αυτό στάδιο και να οδηγήσουν σε μια οργανωμένη και ομαλή μετάβαση την ΑΕΤΟ. Χαίρομαι που από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση του κ. Μόρση θα είναι μια κυβέρνηση που θα εκπροσωπεί πάρα πολλούς τομείς και πάρα πολλά στρώματα στην ε, πολυεδρική και πολύμορφη ε, Αιγυπτιακή κοινωνία. Είναι σημαντικό επίση και να εκπονηθεί ένα νέο σύνταγμα το οποίο θα οδηγήσει σε ένα πολυκομματικό κόμμα που θα σέβεται τι ελευθερίε και τα δικαιώματα και των μειονοτήτων. Έχουν τονίσει και άλλοι ομιλητέ τη σημασία τη κοπτική μειονότητα, τη οποία τα ε, δικαιώματα θα πρέπει να προσπιστούν και θα πρέπει να τύχουν διακρίσεων. Η Αίγυπτος είναι μια κομβική χώρα στον αραβικό κόσμο και σε όλη την περιοχή τη. Ό,τι γίνεται εκεί έχει επιπτώσει σε όλο το μουσουλμανικό κόσμο. Η Αίγυπτος μπορεί να είναι υπόδειγμα, όπω είπε ο πρόεδρο Πέτερινγκ είναι πολύ σημαντικό οι πολιτικοί υπεύθυνοι της Αιγύπτου να καταλάβουν την αναγκαιότητα οι αποφάσεις τους να μην οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση στην περιοχή αυτή η οποία μπαστίζεται από πολλές συγκρούσεις και σειράξεις. Και, ελπίζω ότι θα τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις της Αίγυπτου. Δεν μπορεί να παραμείνει στο περιθώριο η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα τεκτενόμενα με την Αίγυπτο. Είναι μια σημαντική χώρα για την πολιτική γειτονία μα στη Μεσόγειο. Πρέπει να παρακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία προσπαθώντα να υποστηρίξουμε πάντα την υποστήριξη των θεμελιωδών αρχών που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλο, θέλω να υποστηρίξω και το Ίδρυμα Κόνατα Αντενάουερ και να δείξω την αλληλεγγύη με αυτό γιατί περνάει δύσκολε στιγμέ στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ελχάντραουι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Οι τελευταία μήνες ήταν συγκλονιστική στην Αίγυπτο με δράμα, εντάσεις ε, και παράλληλα βεβαίω με την εκλογή Προέδρου είχαμε και συζητήσεις για το νέο σύνταγμα ή δηλαδή τις εξουσίες του νέου Προέδρου και έχουμε άρα ως αποτέλεσμα το ότι κέρδισε αντίπαλο των ενόπλων δυνάμεων αλλά Βεβαίω ε, από ό,τι φαίνεται, κρατάνε ακόμα τα νήματα στα χέρια τους οι στρατιωτικοί. Πρέπει να δούμε τα θετικά αυτών των εξελίξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τώρα την αποστολή να συνεισφέρει στην επιτυχία της δημοκρατικής μετάβασης και ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση θα είναι να σταθεί η χώρα στα πόδια της ε, οικονομικά. Ο τουρισμός έχει καταρρεύσει, εξωτερικές επενδύσεις δεν υπάρχουν, το ταμείο είναι μείον. Οπότε θα πρέπει να συνεισφέρουμε για να ξαναξεκινήσει να λειτουργεί η οικονομία στην Αίγυπτο, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για επιτυχή δημοκρατική μετάβαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ελχαντραουή. Ακολουθεί ο κύριος Κάριμ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρόσφατα επέστρεψα από μία επίσκεψη που έκανα στην Αίγυπτο μαζί με άλλου συναδέλφους ήταν πριν τις προεδρικές εκλογές και ήταν ξεκάθαρο ότι η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη. Γινόταν μάχη εξουσίας μεταξύ το Σύνταγμα μεταξύ των διαφόρων ομάδων και δημιουργούταν το κοινοβούλιο σε αυτή την φάση, οπότε είχαμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή και να μιλήσουμε τα εκλεγμένα μέλη όταν ήμασταν ακόμα εκεί και θα πρέπει να σας πω κύριε Πρόεδρε, ότι δεν είχα μεγάλη εμπιστοσύνη ότι εκείνα τα μέλη θα οδηγούσαν σε ένα πρόγραμμα ανοιχτή προσέγγιση και φιλελευθερωποίηση. Έχω πραγματικέ ανησυχίε για τα δικαιώματα θρησκευτικών μειονοτήτων και των γυναικών. Αλλά ποιο είναι το πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξει την Αίγυπτο που έχουμε μπροστά μα σήμερα. Θα πρέπει να την υποστηρίξουμε, αλλά όχι με έναν τρόπο που εκείνοι που έχουν την εξουσία να μπορούν να ακυρώνουν και να ξεβετερώνουν εκείνους που έχουν διαφορετική άποψη. Η υποστήριξή μας θα πρέπει να είναι προς εκείνους τους ερετούς εκλεγμένους που θέλουν να δημιουργήσουν μια κοινωνία που εδράζεται επί θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επί κοινών αξιών. Ο κ. Πέτερινγκ μιλά ως χριστιανός. Εγώ απαντώ ως μουσουλμάνος. Μιλάμε την ίδια γλώσσα. Ε, είμαστε μια ανθρωπότητα και αυτό θα πρέπει να το εντάξουμε στην κοινωνία της Αιγύπτου που αναπτύσσεται σήμερα στον ιστό της. Ευχαριστώ κύριε Καρίν. Ο κύριος Βίγκενίν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευθύ εξ αρχή ξέραμε ότι η μετάβαση τη Αιγύπτου θα ήταν μακρά, ε, με σκαμπανεβάσματα. Έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε για την Αίγυπτο. Θεσμική αβεβαιότητα, οικονομική, κοινωνική κρίση, συνεχώ έλεγχο πλευρά στρατιωτικών και ισχυρή υποστήριξη για τα Ισλαμιστικά κόμματα, τα μετριοπαθή και τα λιγότερα μετριοπαθή. Παρά τι δυσκολίε, οι προεδρικέ εκλογέ διεξήχθησαν με έναν αποδεκτό τρόπο και οργανώθηκαν αυτόν τον τρόπο. Έδειξαν ότι οι κοσμικέ μετριοπαθεί δημοκρατικέ ε, ε, κόμματα ε, επικρατούν στη χώρα. Το κακό ήταν ότι είχαν διαιρεθεί σε πολλού υποψηφίου και τα κόμματα έμαθαν το μάθημά του. Ο νέο πρόσωπο, ο κ. Μορσή, φαίνεται ένα αξιόπιστο άτομο που κατανοεί τι τις τεράστιες που έχει να κρατήσει ενωμένη τη χώρα, να προστατεύσει τις μειονότητες και να εξασφαλίσει ειρηνική συνέχιση της μεταβατικής διαδικασίας στην Αίγυπτο. Ζητώ να του δούμε μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε ότι είναι ένα στοιχείο σταθερότητα στη χώρα, και ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα πρώτα βήματα που κάνει, που υπόσχονται κάποια πράγματα. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε επί των νέων κοινοβουλευτικών εκλογών, να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε τα διάφορα κοσμικά και φιλελεύθερα κόμματα για να μην έχουμε μια συντριπτική νίκη των Ισλαμιστών, κυρίω ε, τον κάδο των Σαλάφη. Και μετά θα πρέπει να ενισχύσουμε τις πιέσεις επί του Ανώτατου Συμβουλίου των Ενόπλων Δυνάμεων ούτω ώστε να ετοιμάσουν την έξοδό του από την εξουσία. Η εξουσία θα πρέπει να είναι στα χέρια του λαού και αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχο που πρέπει να πετύχουμε μαζί. Το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η νέα πολιτική μα αναθεωρημένη τη γειτονία θα πρέπει να έχει σαν στόχο την υποστήριξη μετάβαση για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη τη χώρα και δεν θα πρέπει να αποσπάτει η προσοχή μα στο γεγονό ότι τώρα ο πρόεδρο τη χώρα αντιπροσωπεύει του αδελφού μουσουλμάνου. Θα πρέπει να τον κρίνουμε αυτόν και οδήποτε πολιτικό κόμμα στην εξουσία από τι πράξει του και όχι από τι προσδοκίε μα και το πολιτικό του υπόβαθρο και την ιστορία του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Ερχόμαστε τώρα στη διαδικασία οφθαλμοθυρίας και θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Χάουιτ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που μπορώ να συμβάλλω σε αυτή τη συζήτηση. Πολλοί από εμά φοβούνται ότι καθυστέρηση της ε, ανακοίνωσης των ε, αποτελεσμάτων στην Αίγυπτο ε, κάλυπταν κάποια χειραγώγηση της ψήφου και θα ήθελα να πω στους συναδέλφους στην στη συζήτηση ότι είναι παράξενο ε, τελικά που έγινε μια μετάβαση σε αυτή τη χώρα και αυτό είναι κάτι ευπρόσδεκτο χωρίς να εγκρίνουμε συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Υπήρχε η προπτική όλη η Αραβική Άνοιξη να σταματήσει εάν αυτές οι εκλογές είχαν αποτύχει. Και πιστεύω ότι απομένουν κάποιες ελπίδες με αυτά που συνέβησαν στην Αίγυπτο. Ε, συνάντησα εκπροσώπου των αδελφών μουσουλμάνων στο Κάιρο μαζί με άλλου συναδέλφου. Μα είπαν ότι θέλουν πλουραλιστική δημοκρατία, δικαιώματα των μειονοτήτων, δικαιώματα των γυναικών. Δεν πρέπει να είμαστε επιθετικοί. Ακούμε κάτι, ε, επιθετικές θέσεις κατά του πολιτικού Ισλάμ από την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να είμαστε και αφελεί όμω, Αλλά θα πρέπει να του δείξουμε εμπιστοσύνη για τι υποσχέσει που έδωσαν. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Αραβική Άνοιξη και τις αλλαγές που γίνονται στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και η κυρία Σαγκεντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα αίτημα προς εσάς. Ε, είδαμε τις εκλογές στην Αίγυπτο και είχαμε πράγμα τον πρώτο ελεύθερα εκλεγμένο πρόεδρο τον κύριο Μόρση αλλά πριν μπορέσει να ξεκινήσει ήδη ο στρατός του αφαίρεσε κάποιες αρμοδιότητες και θα ήθελα να προτείνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βιαστεί να προσκαλέσει τον Πρόεδρο να έρθει εδώ πέρα να μας μιλήσει και να στείλει το μήνυμα άρα στην Αίγυπτο πως μιλάμε με ε, ελεύθερα εκλεγμένους εκπροσώπους του λαού και προέδρους και πώς τον βλέπουμε αυτόν ως συνομιλητή μας και όχι τον στρατό. Αυτή είναι η παράκλησή μου προς εσάς και θεωρώ πως εάν γίνει κάτι τέτοιο θα έχουμε κάνει νομίζω θα έχουμε περιβήσει μεγάλη τιμή στον Αιγυπτιακό λαό και στον Αιγύπτιο πρόεδρο. Σας ευχαριστώ κυρία Σαρκεντίνη. Ογκριώθηκε η διαδικασία και τον λόγο έχει ο κύριος Μαυρογιάννης για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω μόνο λίγα λόγια για κάποιες από τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει από τα διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχήν για την καταπίεση των ΜΚΟ που έχουν εξωτερική υποστήριξη. Αυτό είναι κάτι που μας οδηγεί σε μεγάλη ανησυχία. Η ΜΚΟ είναι σημαντικό στοιχείο δημοκρατικών κοινωνιών. Η υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να είναι και ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής μας γειτονία. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει παρακολουθήσει το θέμα αυτό πολύ προσεκτικά. Η υπάτη εκπρόσωπος, κυρία Άστον, έχει εκφράσει τις ανησυχίες της για τους περιορισμούς στην οργανώση της κοινωνίας των πολιτών με δύο δηλώσεις ενώπιον και του Κοινοβουλίου αυτού. Το θέμα αυτό επίσης έχει αντιμετωπιστεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών 20 Φεβρουαρίου 2012. Επίσης, όταν υπάρχουν διώξεις εναντίον Απασχολούμενο από μη αυτό είναι κάτι το οποίο δείξε σε αντίδραση της κυρίας Άστος στις 21 Φεβρουαρίου 2012 όταν τονίσαμε τις ανησυχίες μας και ζητήσαμε να υπάρξει αναβολή αυτών των ε, ερευνών μέχρι να υπάρχει νέα νομοθεσία για τις ΜΚΟ. Όπως ξέρετε έχει αναβληθεί αυτή η δικαστική διαδικασία μέχρι τον Ιανουάριο του 2013 και έχουν αρθεί οι περιορισμοί προς τη ΜΚΟ, αλλά οι εκκλησίες δεν καλύπτονται από αυτήν ναι. την ε, ε, ρύθμιση. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να αποδίδει τη μεγαλύτερη δυνατή σημασία στο θέμα αυτό και θα διατηρήσουμε στενές επαφές με την ε, Αιγυπτιακή κυβέρνηση και με τους εταίρους μας και τους Αμερικανούς για να επιληθεί το πρόβλημα αυτό. Κάποιοι από εσά επίσης υπογράμμισαν τη σημασία του να διατηρηθούν οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου. Παρακολουθούμε από πολύ κοντά το θέμα αυτό. Όπως ξέρετε όμως, ο νέος Αιγύπτιος πρόεδρος είπε ότι, και το υπεγράμμισε αυτό, ήταν ιδιαίτερα σαφής, ότι θα τηρήσει αυτές τις συμφωνίες. Θα πρέπει να παραμείνουμε επάγρυπνοι, πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε τη σημασία της δήλωσης αυτής. Θα ήθελα εν τέλει να ευχαριστήσω τα έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καρποφόρα αυτή ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αίγυπτος μετά από την εκλογή του Προέδρου Μόρση. Στα πλαίσια αυτά, οι επικείμενες εξελίξεις μετά από την ε, τροποποίηση του συζητάγματος από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων θα είναι κάτι που θα παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά. Όπως και εσείς πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να διαδραματίσει ένα ιδιαίτερο ρόλο για να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο. Από αυτή την έποψη η Αίγυπτος είναι μια υποδειγματική περίπτωση. Θα πρέπει να επιτύχουμε στον δυνατόν περισσότερα για να υποστηριχθεί η δημοκρατική μετάβαση και τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες στη χώρα αυτή θα πρέπει να συνεχίσουν να την χάνουν προσεκτικής αξιολόγηση. Και στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε και ο πρόεδρος Πέτρινγκ, ορθώς και θέλω να σας αναφέρω τον σεβασμό μου, τον ε, σεβασμό μου προς εσάς κύριε Πέτριν. Πράγματι προσπαθούμε να δούμε Προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη λοιπόν όλα αυτά που είπατε, γιατί σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει η ύψιστη προσοχή που θα αποδοθεί στην θρησκευτική ελευθερία και δεν παραγνωρίζουμε και τα δικαιώματα των γυναικών στην Αίγυπτο, εξ ονόματος της κυρίας Άστον, της ΥΠΑ του εκπροσώπου και αντιπροέδρου, σας διαβεβαιώνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να αποδίδει τη μεγαλύτερη σημασία στην Αίγυπτο. Προσβλέπουμε σε επικοδομητική συνεργασία με τον νέο πρόεδρο και την κυβέρνησή του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μαυρογιάννη. Η συζήτηση λοιπόν για την Αίγυπτο έχει τελειώσει. Η επόμενη συνεδρία σε Ολομέλειας είναι αύριο από τις 9 έως τις 2 και από τις 13 μέχρι τις 19 έχει εξαντληθεί η ημερήσια διάταξη και θα είναι η ημερήσια διάταξη θα είναι